Πρόεδρε, συγγνώμη. Είναι ένα διαδικαστικό κάτι που έξω συνέβη πριν λίγο. Βγήκα και είδα ήδη από το πρωί ένα βλάσφημο πίνακα κατά την άποψή μου. Ένας ε, Χριστός με δίπλα, ε, γονατιστός και δίπλα του μια γυμνή γυναίκα. Ζήτησε να φύγει ο πίνακας αυτός, δεν πήρα απάντηση, πήρα τον πίνακα, τον έβγαλα εγώ όταν, ε, για να τον ε, δώσω στους αρμόδιους, μετά πήγα κάπου αλλού και με σταμάτησε κάποιος της ασφάλειας, με αντιμετώπισε σαν εγκληματία. Ε, πριν σε ένα μήνα θα έρθει ο, ο Πάπας. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιους βλάσφημους πίνακες ε, εδώ. Όποιοι είναι καθολική όπω εγώ πρέπει να αισθάνεται κάθε φορά που μπαίνει προσβεβλημένο βλέποντα τέτοια πράγματα. Αν βγω και ξαναδώ τον πίνακα αυτό θα μου έρθει ξανά η βούληση να τον αφαιρέσω. Η θρησκεία μου επιβάλλει, η, η άρνηση τη θρησκεία μου επιβάλλει να δω κάτι που δεν δέχονται. Πώ μπορώ να δεχθώ άλλε θρησκείε, ρωτώ. Αν ήταν έξω ο Μωάμεθ και δίπλα του μια γυμνή γυναίκα κάποιο θα έλεγε κάτι. Η χριστιανική θρησκεία, ο καθολικισμός, δεν μπορούν να συνεχίσουν να βλέπουν τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να πω γιατί πραγματικά αισθάνθηκα ότι με αντιμετώπισε σαν εγκληματία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πρόεδρε. Απλά ήθελα να πιστήσω την προσοχή σε αυτό. Με περιμένουν απ' έξω να με πιάσουν η ασφάλεια. Κοιτάξτε, έχετε ένα λεπτό για μια διαδικαστική παρέμβαση. Και ήταν σαφές ε, περί τίνος επρόκειτο. Θέλω να σας προτείνω το εξής. Εάν θεωρείτε ότι έχετε προσβληθεί, από τα κτίρια, από, τα, από το έργο αυτό τέχνης να ζητήσετε να ελεγχθεί από τον αρμόδιο κοσμητό